Der Präsident. Ich Επαναλαμβάνει τη συνεδρίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα έχουμε μια διαδικαστική πρόταση από τον κύριο Αουστρεβίτσιους. Κύριε Αουστρεβίτσιους, έχετε το λόγο. Mr. Κύριε Πρόεδρε.